Ταμείο Αφετηρία τη επίλυση των διαφορών στον ΠΟΕ όπου ανήκει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ολοκλήρωση της συζήτηση. έχουμε πρόταση ψηφίσματο, η οποία θα ψηφιστεί αύριο το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ και τώρα έχουμε μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία εμβολίου κατά της φυματίωσης από την ομάδα των φιλελευθέρων και άλλους συντάκτες. Κύριο Γκέρεν, εκ μέρου των για πέντε λεπτά. Κύριε Γκέρεντ, έχετε την καλοσύνη να λάβετε το λόγο για πέντε λεπτά. Θέλετε. Κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, θέλετε το λόγο. Είστε συντάκτη. Τη προφορική ερώτηση προτιμάτε όχι. Τρεις φορές προσπάθησα να σας καλέσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Ήσταν απασχολημένος με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Με πολύ μεγάλη χαρά θα προσφέρω την υποστήριξή μου σε ένα πανευρωπαϊκό εγχείρημα, πολύ φιλόδοξο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα αναπτυσσόμενα κράτη, που στόχο έχει να θέσει τέρμα στην επέκταση της σηματίωσης, δηλαδή να εξασφαλίσει την, εκρίζωση, την εξάλληψή της χάρη στην, ε, στον εμβολιασμό. Μην ξεχνάμε ότι περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο έχασαν ε, τη ζωή του 2009 λόγω της φυματίωσης, δηλαδή 4.700 άτομα καθημέραν και μην ξεχνάμε και πόσο μεγάλο οικονομικό κόστος μπορεί να έχει αυτό, πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο μόνο για την Αφρική. Άρα η φυματίωση δεν μπορεί να αναχθεί μόνο σε ε, πρόβλημα των αναψωμένων κρατών. Θα ήταν εσφάλμα κάτι τέτοιο. Και σημειώνουμε ότι τα κρούσματα φυματίωσης που καταγράφηκαν το 2009 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία μας υπενθυμίζουν πόσες ε, καταστροφές μπορεί να επιφέρει αυτή η αρρώστια που εκτείνεται και στις δικές μας χώρες ε, στην Δυτική Ευρώπη αλλά και στα ανατολικά μας, στην Ελλάδα, τη Μολδαβία και τη Ρωσία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειε για την ανάπτυξη αποτελεσματικών ε, εμβολίων, ιδιαίτερα για τι αναπτυσσόμενε χώρε και σε τιμέ ανεκτέ. Δεν θέλω να πρέπει να επισημάνω τα εξή. Καταρχά ότι, ότι η υγεία δεν έχει τιμή, αλλά έχει κόστο. Έχει μου η ικανότητα των ε, πληρωμών ε, παραμένει περιορισμένη στις βιομηχανοποιημένες χώρες ε, και πρέπει να γίνει κατανομή του άχθους. Οι ασθενείς του Βορρά των βιομηχανοποιημένων χωρών θα πρέπει να πληρώσουν ισχυρό τιμήμα αν οι πόροι της έρευνας δεν αυξηθούν γρήγορα και η χρηματοδότηση των χωρών του Νότου παραμένει αναπαρκής και μάλιστα θα είναι και σχεδόν συμβολική. Έτσι λοιπόν πρέπει εμείς να είμαστε λέγια για να καλύψουμε αυτή την ανεπάρκεια. Δεύτερο σχόλιο, η πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης λαμβάνει τη θέση της στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και απεικονίζει ε, γιατί μπορούμε να πράξουμε αν εγκαίρως μπορέσουμε να χαράξουμε προτεραιότητες στον τομέα της υγείας. Και τρίτο σχόλιο, και θέλω να ολοκληρώσω με αυτό, ε, τίποτα δεν αποκλεί την πρόσθετη χρηματοδότηση, ε, όπως το χάρη από διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλα κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς ε, ή πολλές αναδυόμενες χώρες που θίγονται από το πρόβλημα της σηματίωσης, είτε άμεσα σε επίπεδο πληθυσμού είτε έμεσα λόγω της διεθνούς αλληλεγγύης θα έπρεπε ε, λογικά να συνεισφέρουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Πρόκειται ε, για την ε, εταιρική σχέση δημόσιο και ιδιωτικού τομέα και αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να φέρει την αλληλεγγύη σε αυτούς που έχουν ιατρικές και οικονομικές ανάγκες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για να απαντήσει τώρα, παρακαλώ τον λόγο, λόγο κύριος Επίτροπος. Κύριε Τσόλος. Το 2008 η πρωτοβουλία αυτή για το εμβόλιο καταστηματίωσης ήταν οργάνωση ιδιωτική και στα πλαίσια του οδό προγράμματος πλαισίου για την ε, έρευνα κινητοποίηση επιπλέον ε, πόρους γιατί ήταν θεοσοβρό το θέμα και τότε είχαμε ε, κάποια εμβόλια τα οποία ακόμα βρίσκονται σε, σε πρόορη φάση ανάπτυξης και τονίστηκε το ότι δεν έχουμε κλινικά δεδομένα ούτως ώστε να θεωρείται βάσιμη ιδέα το ότι ένα από τα αναπτυσσόμενα υποψήφια εμβόλια θα μπορούσε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό από αυτό το οποίο χρησιμοποιείται τώρα αυτός ο Βάκυλος Γκέρεν και θα πρέπει για να μπουν στην αγορά τα καινούργια εμβόλια να αποδείξουν ότι έχουν ε, ε, αποτελεσματικότητα σε σχέση με αυτό τον παραδοσιακό βάκελο ή να είναι ακόμα καλύτερα και να εκτοπίσουν, να αντικαταστήσουν αυτό το παραδοσιακό. Θέμα ότι δεν έχουμε πάντοτε, ακόμα δεν έχουμε αυτού του είδους τα, τα δεδομένα. Οπότε αυτή η πρωτοβουλία βολή του κατά δεν θεωρείται απομονωμένη σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες τόσο ώστε να μπορέσουμε τις κλινικές δοκιμές να τις υποστηρίξουμε οπότε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Αυτή η, αυτός ο ευρωπαϊκός φορέας ανέλαβε την πρωτοβουλία δυνάμει του άρθρου 185 σύμφωνα με το οποίο έχουμε 14 κρατημέλη και δύο συνδυομένες χώρες αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλοι μαζί δεσμεύτηκαν ε, 85 εκατομμύρια ούτως ώστε να γίνει αυτή η έρευνα για εμβόλια, για ελονοσία, AIDS, ε, φυματίωση στις χώρες κάτω από τη νοτίου της Σαχάρας, ούτως ώστε μέχρι το 2015 είπαμε θα ε, ολοκληρώνουν τις σχετικές δοκιμές και επίσης αυτές που αφορούν το εμβόλιο για την φυματίωση, οπότε έχουμε και εναλλακτική που ήδη τρέχει. Ε, εμείς μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε αυτό που ονομάζεται πρότυπο επιχειρηματικό από συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού αλλά επίσης και το μοντέλο της πρωτοβουλία εμβολίου για τις Και θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ σημαντικό όργανο πολιτικής στο μέλλον. Όμως θα πρέπει να έχουμε εις βάθος ανάλυση τη, ε, της εμπορικής όσο και αποτίμηση του κινδύνου. Επομένως, θα προχωρήσουμε έχοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, τόσο ώστε οι δοκιμές να μου αδείξουν κάτι βάσιμο. Ε, επίσης, πρέπει να λυθούν τα μοντέλα σε συνεργασία με τις ε, συνεργασία με τράπεζες και σχετικά ιδρύματα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα έχουμε εφαρμογή στην πράξη της πολιτικής ενόψης του 2020 και για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και τώρα έχουμε τους ομιλητές εκ μέρους των ομάδων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Δημοκρατών, η κυρία Καρβάλιο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τα κρούσματα της φυματίωση σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχίζουν να ε, προκαλούν μεγάλε ανησυχίε παρά την πρόοδο που έχει υλοποιηθεί ε, λόγω στο ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, επιστημονική έρευνα. Λόγω αυτού σήμερα πεθαίνουν δύο εκατομμύρια άτομα λόγω της φυματίωσης μέσω του σημερινού ψηφίσματο και μέσω της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φυματίωσης καλούμε ε, να έχουμε ε, περαιτέρω έρευνες για να αναπτύξουμε εμβόλια κατά αυτής της νόσου τα εμβόλια είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να προστατευτούν οι πολίτες από τις λοιμώδεις νόσους αλλά είναι σημαντικό ε, και να φτάσουν αυτά τα εμβόλια και στις αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να διασωθούν ζωές και να καταπολεμηθεί ανέχεια συνέχεια, όπως ανέφερα, έχουν έχει γίνει κάποια πρόοδο και είμαστε σωστοί εδώ, αλλά πρέπει να αναλάβει νέα δέσμευση Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλέσουμε για μια νέα συντονισμένη δράση και ενίσχυση τη ευρωπαϊκή έρευνα για την καταπολέμηση των όσων που έχουν να κάνουν με τη φτώχεια. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να εξελίψουμε την, και να μειώσουμε αυτή την ε, κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι σε αναπτυσσόμενε χώρε. Ε, πρέπει να ε, γίνουν περαιτέρω προσπάθειες έρευνας σε αυτό το τομέα και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας να μεταφραστούν υπέρ το ωφέλου του πληθυσμού στα πλαίσια τη στρατηγική τη Ευρώπη του 2020. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρου τη ε, ομάδα προοδευτική ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών τη Ευρώπη, ο κ. Κάσμαν, παρακαλώ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με χαρά σα βλέπω πάντα όταν προεδρεύεται σε τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με τα δεινά και την ασθένεια που πλήττει τους ανθρώπους και ξέρω ότι εσείς πάντοτε με κατανόηση παρακολουθείτε τα θέματα αυτά και με συμπόνια. Θα ήθελα λοιπόν να αφαιρθώ και εγώ στο θέμα αυτό της φυματίωσης. Είναι όντως ο δεύτερος, το δεύτερο αίτιο θανάτου από λοιμώδης νόσους. 1,6 έως 2 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στον κόσμο από τη φυματίωση και έχει αναπτυχθεί ένα ε, γερό σχέδιο μια πρόοδο σημαντική ως προς τα εμβόλια κατά τη φυματίωση, όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος, Δυστυχώ όμω τώρα η χρηματοδότηση και στην Ευρώπη και στι αναπτυσσόμενε χώρε ε, δεν δίνουν αρκετό χρόνο και ε, χρηματοδότηση στις φάσεις 2 και 3, δηλαδή τις κλινικές δοκιμές, για να ξέρουμε ότι είναι ασφαλή τα εμβόλια. Εμβόλια υπάρχουν, αλλά πρέπει να είμαστε και βέβαιοι ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά πριν λάβουν την άδεια να χορηγηθούν στους πολίτες. Θα μου πείτε, χρηματοδότηση άλλη δεν έχουμε. Ωραία. Μπορώ τουλάχιστον να ρωτήσω όμως εάν Υπάρχει δυνατότητα από τις σχετικές διατάξεις η χρηματοδότηση να στοχεύει ειδικά τις κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες και η Επιτροπή σκέφτεται την εισαγωγή συμπληρωματικών ε, μηχανισμών χρηματοδότησης για την επιδίωξη της ανάπτυξης ε, νέων ε, και πρωτότυπων εμβολίων για τέτοιες επικίνδυνες και σχετικά σπάνιες αρρώστιες όπως τις φυματίωσης. Ευχαριστώ εκ μέρου των μη εγγεγραμμένων, κυρία Βέρτμαν, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι πολύ δεδομένη ακόμη η φυματίωση κυρίως στα φτωχότερα κράτη. Ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού ε, φέρεται ως φορέα της φυματίωσης και τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο είναι τα θύματα της κάθε χρόνο. Έχουμε 7 θανάτους στην Ευρώπη και ε, 4.900 νέα κρούσματα το χρόνο μόνο στην Ευρώπη. Φαίνεται λοιπόν να περνάει μια περίοδο αναγέννησης η φυματίωση ακόμη και στις χώρες μας. Οι αποτελεσματικοί εμβολιασμοί όμως θα μπορούσαν να περιορίσουν αυτή την πορεία της φυματίωσης και τελικά να βοηθήσουν στην εξάλληψή της. Εάν έχουμε κατάλληλα εμβόλια είναι δυνατή η εξάλληψη. Αυτή τη στιγμή όμως ε, υπάρχουν πολύ ανθεκτικά ε, πολύ ανθεκτικές εκδοχές του, ε, της φυματίωσης και θα πρέπει να κάνουμε τις μελέτες εκείνες που χρειάζονται σε τα ε, εμβόλια που θα αναπτύξουμε είναι αποτελεσματικά και ασφαλή. Ευχαριστώ και τώρα κύριο Κάτσουμερα και για δύο λεπτά. Κυρίες και κύριοι, πριν έρθει η ώρα της εφαρμογής αυτής της πρωτοβουλίας είχαμε σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά ασθενείς, θνησιμότητα και σε Ασία και Νοτιού Σαχάρας παραμένει το πρόβλημα αυτό. Δύο δις υπολογίζεται ότι είναι φορείς αυτού του μικροβακτηρίου, δηλαδή το 1 τρίτον του πληθυσμού της ε, και ένας στους 10 εξ αυτών πρόκειται να ασθενήσει. κυρίως ε, όταν έχουμε άσχημες συνθήκες ε, ε, στέγασης, διαβίωσης, κακή διατροφή, στρες, τότε ευνοείται αυτή η ασθένεια οι κυβερνήσεις στις ανεπτυγμένες χώρες δεν δαπανούν αρκετά σε αυτό το μέτωπο. Άρα η ύπεθρος υποφέρει ακόμη περισσότερο. Δεν υπάρχουν τα μέσα επομένως για καταπολέμηση της ασθενείας. Γι' αυτό και φτωχές χώρες είναι αυτές που περισσότερο πλήσονται και ακόμη περισσότερο σε αυτές τις χώρες η, η Ήπεθρος. Σαν τις χώρες, σαν έχουμε 5% του προπολογισμού και 2,5% στις ε, αναπτυσσόμενες Όμω δεν είναι δυνατόν να δαπανίσουν περισσότερο φτωχέ χώρε, να υπάρξει τοργική βοήθεια, το είπε ο κύριο Γκέρεν, γιατί εδώ πέρα δεν πρόκειται μόνο για μεγάλο ιατρικό πρόβλημα, είναι και κοινωνικό και οικονομικό έχουμε εδώ ως συνέπεια πτώση παραγωγικότητας. Άρα θα πρέπει εμείς άμεσα να κάνουμε κάτι αυτό το πρόβλημα και θα πρέπει αυτά τα εμβόλια να είναι σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ λίγο Πρόεδρο. Ευχαριστώ Κορτές Λάστρα δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η υγεία είναι κάτι που μας απομένει για την καταπολέμηση της στόχιας να καταρχήν πρέπει να καταπολεμήσουμε την παιδική τα δεύτερον να βελτιώσουμε την υγεία των μητέρων να καταπολεμήσουμε την ελληνοσία το AIDS και πετώλας ένας νόσους μεταξύ των οποίων και η φυματίωση παρόλα αυτά όλοι είμαστε παρόντες εδώ γνωρίζουμε ότι οι στόχοι αυτή της κλητίας ε, είναι οι πιο καθυστερημένοι αυτή τη στιγμή. Ε, πρέπει να λάβουμε μέτρα και να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για τα προγράμματα υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες η πρόσβαση σε δωρεάν συστήματα περίθαλψης πρέπει να είναι ε, τελικό στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα. Πρέπει να υποστηρίξουμε ε, τα ταμεία ενίσχυσης για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης, της ελληνοσίας, αλλά είναι και απαραίτητο να υποστηρίξουμε πολιτικά και οικονομικά τις χώρες αυτές για να μπορέσουν να αναπτύξουν συστήματα υγείας αποτελεσματικά. Είμαι σίγουρος ότι αυτή θα ήταν, αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να διασφαλίσουμε ε, την αρχή του ownership και να επιτρέψουμε την πρόσβαση του πλέον ωφελού του πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σαμπόρσκα. Παρακαλώ δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η είναι μια πανδημία μαζί με την ολονοσία για το έτσι πιο σημαντικές που έχουν τόσο σοβαρές επιπτώσεις για Ασία, Αφρική, τις αμπισόμενες εκεί χώρες εκεί έχουμε ως ε, επιπτώσεις πάρα πολλές σοβαρές οικονομικές ε, επίσης συνέπειες όμως και άλλες χώρες πλήσονται από αυτές τις ασθένειες άρα δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι πρόκειται μόνο για ιατρικό πρόβλημα είναι πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την νοοτροπία, τη συμπεριφορά της ανθρωπότητας γιατί εδώ πέρα επιβάλλεται να υπάρχει αλληλεγγύη, χρειάζεται παγκόσμια αντιμετώπιση. Αυτοί που σαν χώρε χώρες έχουν θύματα αυτής της ασθενείας το παθαίνουν διότι δεν έχουν ικανή ιατρική κάλυψη που θα πρέπει να ερευνήσουμε, να επενδύσουμε, να βρούμε νέα εμβόλια που να αντιμετωπίσουν τις νέες μορφές μεταλλάξεις του προβλήμα της ασθένεια. και επίση τώρα θα πρέπει να πούμε ένα μπράβο στους ήρωες εκείνες που δίνουν τη μάχη τους κατά τις ε, κάθε μέρα αλλά για να μπορέσουν να δώσουν αυτή την, επιτυχία εναντίον αυτών των ασθενειών και αυτών των βακτηρίων κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας και να δώσουμε χέρι βοηθείας στο ιατρικό προσωπικό, στις χώρες εκείνες, γιατί εκεί έχουμε εκροή, φυγή αυτού του προσωπικού, μια που δεν υπάρχει οικονομική κάλυψη, συνέχεια συρρυκνώνεται. Επομένως θα πρέπει για παγκόσμιο πρόβλημα να έχουμε και παγκόσμια ανταπόκριση και πέραν της έρευνας και των φαρμάκων να προσέξουμε και άλλου είδους αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Ευχαριστώ. Έχουμε τη διαδικασία καρσιά τώρα. Ο κύριος Νικολάζητσου πρώτα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να υπογραμμίσω πως η φυματίωση δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί από προσωπουγής και βλέπουμε ότι δύο εκατομμύρια τουλάχιστον το χρόνο είναι τα θύματα αυτής της αρρώστιας. Και θέλω να πω ότι είναι τουλάχιστον θετικό το ότι αναγνωρίστηκε αυτή η σημασία αυτής της αρρώστιας. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία της Επιτροπής, διότι μιλάμε για το AIDS ως πανδημία, αλλά καλό να μιλάμε και για τη φυματίωση, η οποία προξενεί το θάνατο πολλών ανθρώπων στον κόσμο, περί τα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την έρευνα ώστε να φτάσουμε σε νέα εμβόλια. Πολύ σωστά. Είπε όμως και η Επιτροπή ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα εμβόλια. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή, στα στάδια πρώτης κλινικής δοκιμής. Και πρέπει να δοκιμαστεί ακόμη η αποτελεσματικότητά του σε πραγματικές συνθήκες. Ολοκληρώνω, Πρόεδρε. Θα ήθελα πιο πολλά κονδύλια για την έρευνα να ζητήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η θενσιμότητα πάει από το 1,6 μέχρι 2 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως και γι' αυτό είναι αυτή η ασθένεια ε, μία από τις βασικές αιτίε ε, θανάτου από μοσμετικές ασθένειες και γι' αυτό και ανησυχούν οι οργανώσεις υγείας. Έχει προοδεύσει σήμερα η ιατρική. Όμως θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι ήρθε η ώρα να αντικαταστήσουμε το κλασικό εμβόλιο με άλλο, πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε από τη μια μεριά πιο γενναιόδορη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα. Όμω από την άλλη μεριά χρειάζονται και νέοι τρόποι χρηματοδότηση όπως ε, αυτό, αυτή η πρωτοβουλία η οποία κατευθύνεται προς καινούριε εναλλακτικέ για έτσι να έχουμε ε, και ελκυστικότερη κατάσταση για τις ε, επιχειρήσεις οι οποίες να βάλουν και αυτές το δεθαράκι και να στηρίξουν. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Η φυματίωση πριν από ένα περίπου αιώνα μάστιζε την ε, Ιρλανδία, την πατρίδα μου, προξενούσε πολλούς θανάτους. Μπόρεσε για 36 χρόνια σχεδόν να εξαφανιστεί, αλλά δυστυχώς, όπως υπόθηκε νωρίτερα, επανεμφανίζεται και είχαμε θύματα ένα παιδί και ένα βρέφος πέρυσι. Δύο εκατομμύρια ανθρώπων που αρρωσταίνουν από το βακτηρίδιο αυτό και τα θύματα που θρυνούμε κάθε μέρα πρέπει να μας πείσουν να βοηθήσουμε για περισσότερη έρευνα σε αυτή την ε, ε αντιμετώπιση της φυματίωσης. Πέραν της, ε, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας έχουμε ηγετική θέση στην έρευνα για τα εμβόλια και των δύο τύπων του βακτηριδίου. Ο κύριο Φεραίρα, ευχαριστώ. Τέσσερα έτη έχουν απομείνει για την υλοποίηση των στόχων τη χιλιετία και τέσσερα χρόνια πριν η φήματίωση. παίρνει δύο εκατομμύρια ζωής το χρόνο. Ναι, έτσι λοιπόν γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ε, μία ε, νόσο που δεν συναντάται ιδιαίτερα στι βιομηχανικέ χώρε. Το πρόβλημα τη φηματίωση όπω και νόσων δεν ε, επιλύονται αν δεν υπάρχουν ποιοτικέ υπηρεσίε υγεία όπου έχουν πρόβλημα πρόσβαση ε, όλοι οι πολίτες, η πολιτική συνεργασία και αναπτυξιακή ε, ε, συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνει και ανάπτυξη προγραμμάτων εμβολιασμού αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και μηχανισμοί χρηματοδότησης που να επιτρέπουν να θέσουμε τέλος σε καταστάσεις εξαθλίωσης και υποδούλωσης στον τρίτο κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα ο κύριος Τσέκετη, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, η Ουγγαρία γνώρισε τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων προξενή η φυματίωση. Αυτό οφείλεται σε μια ε, αυτό μάλλον οδήγησε σε μια ε, διαφορετική θεώρηση της κατάστασης και την εισαγωγή νόμου το 2006 για καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας. Το ίδιο βλέπουμε και σε ε, και, γενικότερα προς την αντιμετώπιση τις φυματίες αλλά και τη διάγνωση και τα προληπτικά εμβόλια και τη δυνατότητα εξασφάλιση αυτών των εμβολίων για οποιονδήποτε βρίσκεται σε ένδια και τα χρειάζεται. Έτσι μπορούμε να έχουμε έθνος, Ευρώπη και κοινωνία πολύ πιο υγιή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για να κλείσει τη συζήτηση θα λάβει το λόγο ο Επίτροπος κ. Τσόλος. Ευχαριστώ. Θα ε, προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις όσες ακούστηκαν. Καταρχήν, ε, πράγματι υπάρχει ανάγκη να γίνουν περαιτέρω έρευνες, ε, όπως είπα και στην εισαγωγή μου η Κομισιόν να ε, αναζητεί οδούς για να τροφοδοτήσει ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα ε, για τη φυματίωση. Μία λύση θα μπορούσε να είναι η ανανέωση του προγράμματος ε, το οποίο, για τον οποίο σας μίλησα, το οποίο ε, λειτουργεί τώρα με 400 εκατομμύρια ευρώ, 200 εκατομμύρια από την Κομισιόν. Η Κομισιόν σκέφτεται και την δυνατότητα να έχουμε και τη συνέχεια του προγράμματος, αν είστε 2 και πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν ήδη χρηματοδοτεί ε, προγράμματα ερευνητικά για τη φυματίωση. 55 εκατομμύρια ευρώ ήδη χρησιμοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση, αλλά είναι αλήθεια ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Η ΕΣΔΙΤ ε, επίσης ε, είναι ένα θέμα προς μελέτη όμως, σε ό,τι αφορά τις διάφορους υποψηφίου ε, για τα εμβολία για να μπορέσουμε να πληρώσουμε ε, κάποιους υποψηφίους ε, για τον εμβολιασμό στα κλινικά στάδια, πρέπει να το δούμε αυτό. Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι μια συνεχιστική μεταδότηση θα μπορούσε να οδηγήσει ε, σε ένα θετικό αποτέλεσμα για τις βιταμίνες ε, και αυτή είναι μια προσέγγιση προς διερεύνηση αλλά τι πρέπει να αποφύγουμε να αποφύγουμε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Ε, έτσι λοιπόν είναι μια προς μελέτη, αλλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Τώρα, μιλώντας ε, πιο γενικά για τα συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ε, και στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία, αυτό είναι ένα στόχο μέσα και στα, ε, μάλλον και των διάφορων προγραμμάτων που προσπαθεί να ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμοστούν στα διάφορα κρατημέλη. Προσπαθεί να τα κρατημέλη να επενδύσουν στην υγεία στο πλαίσιο τη έρευνα μία από τις πρωτοβουλίες έρευνας και κοινοτομίας ή κομισιόν, μία ομάδα επιτρόπων εργάζεται από αυτού, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να δώσουν όθηση στην καινοτομία για να υπάρχουν περαιτέρω έρευνες και στον τομέα της υγείας, παράλληλα με ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη γέννηση του πληθυσμού. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη πράττει πολλά με το Ταμείο Ανάπτυξης, στον τομέα της υγείας. Δίνουμε έμφαση και φυσικά η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα αυτό. Εξ ονόματος της Κομισιόν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι ανησυχίες σας σε αυτό το τομέα είναι και ανησυχία της Κομισιόν και αφορούν τον τομέα της έρευνας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ προβλέπονται έτοιμα ε, πρόταση ψηφίσματος των φιλευθέρων, των πρασίνων, των, ε, της ΓΚΟΕ.